Στη συνέχεια έχουμε τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής σε σχέση με την έκβαση της Συνόδου G20. Ο κύριος Κότζη έχει το λόγο εξ ονόματος του Συμβουλίου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη δυνατότητα που δίνετε στην Προεδρία και ειδικά στην Ιταλία που είναι μέλος των G20 να ε, ανοίξει τη συζήτηση. Όπως ξέρετε ήταν παρόντες και ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα αποτελέσματα ήταν πολύ θετικά διότι σχετίζονται με τις θέσεις μας στον οικονομικό τομέα. Προτείναμε κατά το εξάμεινο αυτό το θέμα της ανάπτυξης. Το θέμα της ανάπτυξης ε, εφήγει από όλου στο Brisbane. Δεν το έθιξε μόνο η Ιταλία αλλά και πολλοί άλλοι. Δηλαδή δεν πρέπει να βλέπουμε ε, την ανάπτυξη και τη λιτότητα σαν ένα δίδυμο, θα πρέπει να ασχοληθούμε πολύ περισσότερο με την ανάπτυξη. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο ανέκυψε από τη διάσκεψη των G20. Η οικονομία γνωρίζει ένα επιβραδυμένο ρυθμό σε σχέση με εκείνη της Ιαπωνίας. Είναι ευάλωτη σε παγκόσμιο επίπεδο και δεν μπορεί να δεχτεί άλλους κλειδονισμούς. Και μιλήσαμε και για την πρόοδο που έχει επιτελεστεί. Θα πρέπει να δείξουμε ανθεκτικότητα. Αυτό αφορά ιδιαίτερα το τραπεζικό σύστημα μέσα στα πλαίσια της Τραπεζικής Ένωσης και των τεστ αντοχής τα οποία εκτελούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιες είναι οι συνολικές προτάσεις. Θα πρέπει να προτείνουμε ένα σύνολο στρατηγικών ανάπτυξης με βάση τις δημόσιες και τις ιδιωτικές επενδύσεις, να προωθήσουμε την ανταγωνιστικότητα και να αυξήσουμε το εμπόριο και την απασχόληση. Ιδιαίτερα τη δέσμευσή μας για την αύξηση της ζήτησης μέσω μιας νέας πολιτικής εσωτερικών επενδύσεων και ιδιαίτερα επενδύσεων για να δημιουργήσουμε ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο που περιλαμβάνει και νέα μέσα. ιδιαίτερα υπέρ των ε, ΜΜΕ. Υπάρχει μεγάλο χάσμα μεταξύ επενδύσεων που χρειάζονται σε παγκόσμιο επίπεδο και πραγματικών επενδύσεων. Αυτή τη συζήτηση την είχαμε και σήμερα το πρωί όταν μας παρουσίασε σήμερα το πρωί ο πρόεδρος Γιούνκερ το σχέδιο επενδύσεων. Αυτό εθίγει στο Brisbane και θα δούμε και το Global Infrastructure Initiative. Πέρα από τα τεστ αντοχής και την Τραπεζική Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεισφέρει, όπως τόνισε και ο πρόεδρος της Επιτροπής και όλα τα μέλη των G20 θα πρέπει να προωθήσουμε τις επενδύσεις όπως ε, τις ε, παρουσίασε σήμερα το πρωί ο πρόεδρος Γιούγκερ. Για, για μας είναι μια πρώτη απάντηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε εθνικό. Επίσης, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου Θέλουμε να καταπολεμήσουμε την φοροδιαφυγή και την φοροαποφυγή έτσι ώστε να φορολογούνται τα πραγματικά κέρδη εκεί όπου αποκτώνται. Αυτό τονίστηκε στο ε, ε, Brisbane. Μιλήσαμε ιδιαίτερα για το profit, profit shifting και θα πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στις διάφορες χώρες μέσα στα πλαίσια νομοθετικών διαδικασιών για ανταλλαγή πληροφοριών και ανέκυψε και το θέμα καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής. Αυτό είναι κάτι που έθιξε ιδιαίτερα και η Ιταλική Προεδρία. Θα πρέπει να γίνουν πολλά βήματα προς τα εμπρός. Ένα άλλο θέμα που μας απασχολεί είναι η έλλειψη προόδου των τις δράσεις του Διεθνούς ε, Νομισματικού Ταμείου. Αυτό αποτελεί μεγάλη προτεραιότητα για τους G20 και ζητήθηκε και από τις ΗΠΑ να προβούν στην κύρωση αυτών των ε, μεταρρυθμίσεων μετά το 2010. Τώρα θα δώσουμε συνέχεια σε αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές και θα, πρέπει να προσεγγίσουμε τις οικονομικές μας πολιτικές σε μία περίοδο όπου η Ευρώπη και η Ιαπωνία θα πρέπει να καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες σε σχέση με άλλους εταίρους. Νομίζω ότι θα μπορέσουμε έτσι να βγούμε από την κρίση. Ο κύριος Ντομπρόφσκης έχει το λόγο τώρα. Um, Ευχαριστώ και πάλι. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Χαίρομαι διότι μου δίνετε την ευκαιρία να ενημερώσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την έκβαση της συνόδου του G20 στο Brisbane, όπου μετέβη εγώ προσωπικά μαζί με τον κύριο Γιούγκερ και ε, τον πρόεδρο του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να πω εξ αρχής ότι χαίρομαι ιδιαίτερως με τα αποτελέσματα αυτής της συνάντησης στο Brisbane. Είναι ενθαρρυντικά και φιλόδοξα αποτελέσματα για την παγκόσμια διακυβέρνηση και και πιστεύω ότι συμφωνούν με τους βασικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα ήθελα να τονίσω τέσσερα βασικά σχόλια. Πρώτον για την παγκόσμια οικονομία. Σύμφωνα με την αποστολή και την παράδοση του G20 η κατάσταση της παγκόσμιας οικονομίας ήταν στις πρώτες θέσεις της ημερήσιας διάταξης. Παραμένουμε αισιόδοξοι αλλά και ρεαλιστές. Οι ηγέτες ε, κάλεσαν ε, τις κυβερνήσεις και τις χώρες να υιοθετήσουν ένα σωστό μείγμα πολιτικής με διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και με χρηματοπιστωτική σταθερότητα και ασφάλεια. Αυτοί είναι οι τρεις πυλώνες της οικονομικής μας πολιτικής, άρα συμφωνούμε απολύτως με ε, αυτό. Για ενισχυθεί η ανάκαμψη, η Αυστραλιανή Προεδρία εστίασε το ενδιαφέρον της στα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν για να ενισχυθεί η ανάπτυξη, η απασχόληση, η δημιουργία θέσεων απασχόλησης αλλά και η αύξηση των επενδύσεων. Θα πρέπει να γίνει μεγαλύτερη συσπήρωση για επενδύσεις σε επίπεδο G20, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και λοιπόν ε, μεγάλων χωρών. Επομένως, οι ηγέτες του G20 καλωσορίζουν το πρόγραμμα επενδύσεων 300 δις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ε, σημειώνεται αυτή η πολύ μεγάλη πρωτοβουλία για την κινητοποίηση δημοσίων και ιδιωτικών κονδυλίων για επενδύσεις από το 2015 μέχρι το 2017. Αυτό είναι ένα ισχυρό μήνυμα ενθάρρυνσης ε, στη δική μας επενδυτική πρωτοβουλία και ε, θα πρέπει να ενισχύσουμε τις δράσεις τιτλοποίησης για να συνεχίσουμε να χρηματοδοτούμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεύτερον, ως προς τη διαφάνεια. Οι ηγέτες τόνισαν πόσο σημαντικό είναι να φορολογούνται τα κέρδη εκεί όπου γεννώνται, εκεί όπου δημιουργούνται η φορολογική διαφάνεια είναι κάτι το εξαιρετικά σημαντικό και σε αυτό πράγματι μπορεί να συμβάλλει το G20 και συμφωνούμε απολύτως. Η μεγαλύτερη πρόοδος όμως που έχει σημειωθεί έχει να κάνει με την ε, πρωτοβουλία για το μοίρασμα του κέρδους του ΑΣΑ ε, έτσι ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια, έτσι ώστε να ε, τονιστούν οι αθέμητες φορολογικές πρακτικές διαφόρων χωρών. Δεσμεύθηκαν όλοι να σημειώσουν πρόοδο για όλα αυτά τα θέματα μέχρι το τέλος του 2015. Χάρη στη στήριξη πολλών ηγετών, καταφέραμε στην τελική ανακοίνωση να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα αυτό θα παραμείνει στην ημερήσια διάταξη του G20 όπως και στην ημερήσια διάταξη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από εκεί και πέρα, για το εμπόριο. Λίγες μέρες πριν από τη Σύνοδο ανακοινώθηκε η Συμφωνία Ινδίας Ηνωμένων Πολιτειών για τη διευκόλυνση του εμπορίου και αυτό άλλαξε κάπως το πνεύμα της συζήτησης. και στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της ε, ημερήσιας διάταξης της αναπτυξιακής, αν θέλετε, ατζέντα της ΔΟΧΑ. Πολλές είναι οι προκλήσεις που υψώνονται μπροστά μας και συμφωνήσαμε ότι θα πρέπει το σύστημα να λειτουργήσει καλύτερα εν ώψη της επόμενης συνόδου G20 στην Τουρκία. Τέλος, για τις κλιματικές αλλαγές. Μετά από δύσκολες συζητήσεις, οι βασικοί εταίροι εξέφρασαν τη στήριξή τους, έγινε αναφορά στην κλιματική αλλαγή. Ωστόσο, εμείς δεν μπορέσαμε να δεχθούμε αυτή την ίσονα ε, προσέγγιση. Σε κάθε περίπτωση δουλεύουμε ε, χέρι με χέρι για να προωθήσουμε ακόμα περισσότερο τη θέση μας και καταφέραμε να έχουμε αναφορά στις ε, εθνικές συνεισφορές εν ώψη της COP21 και στο, στο, στην ανάγκη ύπαρξης Ταμείου για το Κλίμα. Έγινε και σχετική συνέντευξη τύπου. Αρχικά πρέπει να σας πω ότι η Αυστραλιανή Προεδρία δεν ήθελε καθόλου να αναφερθεί η κλιματική αλλαγή στο πλαίσιο του G20 και εμείς καταφέραμε αυτό το θέμα και να αναφερθεί και να τονιστεί και στην επίσημη ανακοίνωση, στο επίσημο ανακοινωθέν, αλλά και κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστώ πολύ. Η Πρόεδρος. Σε ευχαριστώ, λέει η πρόεδρο. Τώρα οι ομιλητέ από τι πολιτικέ ομάδες, από το ΕΛΚ. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Μπάλτ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, σα ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σήμερα νομίζω ότι παρουσιάζει, παρουσίασε ένα πολύ φιλόδοξο και απαραίτητο επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη για να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη στην ευρωπαϊκή οικονομία. Καλώ ορίζω ιδιαίτερα το γεγονό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Brisbane ήδη δραστηριοποιήθηκε για το σχέδιο αυτό. Ο κόσμος ε, αναμένει θετικές ειδήσει και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τα κράτη του G20. Αυτές οι δύο πρωτοβουλίες ε, για τις ε, επενδύσεις στα πλαίσια του G20 και στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολλά υποσχόμενες. Να μην ξεχνάμε ότι η αξιοπιστία είναι ο θεμέλιος λίθος της βιώσιμης ανάπτυξης και της απασχόλησης. Υπάρχουν οι ήδη υφιστάμενες δομές οι οποίες θα πρέπει να βρουν συνέχεια και θα πρέπει να παραμείνουν στο σωστό δρόμο. Η φορολογική πολιτική για τις επιχειρήσεις αποτελεί επίσης ένα σημαντικό ζήτημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την ατζέντα του G20. Τα κράτη-μέλη λοιπόν έκαναν ό,τι μπορούσαν για την αυτόματη ανταλλαγή φορολογικών ε, πληροφοριών. Καταλαβαίνουμε βέβαια ότι η κινητήριος μηχανή είναι ακόμα μια πρωτοβουλία του 20 με στενή συνεργασία του ΑΣΑ. Το πρότυπο για την υποβολή αναφοράς είναι κάτι πολύ σημαντικό για τη φορολογία και θα πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει με αμοιβαίο τρόπο και πέρα από το G20. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει η διαφάνεια, η σύγκληση των φορολογικών πολιτικών να συνεχιστεί. Εμείς ως ΕΛΚΑ επιμένουμε στο μέλλον να υπάρχει το εκτεταμένο καθεστώς φορολογίας προκειμένου να υπάρχει και γρήγορο input. Η έκθεση αυτή θα πρέπει να προετοιμαστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα πρέπει να υπάρχει συντονισμός της ε, διαφάνειας και σύγκληση της ε, φορολογικής πολιτικής. Θα πρέπει να συνεχιστούν οι εργασίες και στο πλαίσιο του G20 προς την κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος, για την παρέμβασή σας. Τώρα για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες το λόγο έχει ο κύριος Σίμων. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε να ευχαριστήσω την Προεδρία ιδιαίτερως για την παρέμβαση, για την ε, φοροαποφυγή και για τα επιθετικά σχέδια φορολογίας. Γιατί οι φορολογικές πρακτικές οι οποίες συζητούνται έντονα τελευταία, τις τελευταίες ε, εβδομάδες αποτελούν μόνο την κορυφή του παγόβουνου. Χίλια δισεκατομμύρια υπολογίζεται ότι χάνονται κάθε χρόνο για την φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή. Μιλάμε για οκταπλάσιο. Το τριπλάσιο από αυτό που μας ε, ανέφερε σήμερα ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το επενδυτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι λοιπόν πραγματικά κατεπήγον να δράσουμε και θα πρέπει ως πρωτοπόρος να ηγηθεί των προσπάθειών αυτών η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι ένα πρώτο βήμα, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο όντως θα πρέπει να συνεχίσουμε τη δράση μας. Σωστά λοιπόν τέθηκε το θέμα της φορολογίας στα πλαίσια της ατζέντα του G20 σε ό,τι αφορά ε, μια δίκαιη συμφωνία φορολογίας. Είναι ένα πρώτο βήμα αυτό. Θα πρέπει να ακολουθήσουν και άλλα βήματα όμως. Καταρχάς ε, η πρωτοβουλία του άσα για την μετατόπιση, κατάσταση κέρδους και αποφυγή στην Ευρώπη και σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα πρέπει να τεθεί στο στόχαστρο. Θα πρέπει να φορολογούνται τα κέρδη εκεί που πραγματοποιούνται. Δεν μπορούν να υπάρχουν ε, ε, γελία χαμηλά τέλη για τις άδειες και να χάνονται μεγάλα φορολογικά ποσά σε φορολογικούς παραδείσους. Κατά δεύτερον, χρειάζεται ε, συντονισμένη δράση κατά των φορολογικών παραδείσων. Δεν φτάνει ο ορισμός του ΆΣΑ. Χρειάζεται λοιπόν σαφής ορισμός των φορολογικών ε, οάσεων προκειμένου να τις καταβολευήσουμε. Εμείς προτείνουμε την ε, σύσταση ενός, μιας μαύρης λίστας. Κατά τρίτον, κατά πολέμηση του ξεπλήματος βρώμικου χρήματος οι εταιρείε γραμματοκιβωτίου θα πρέπει να μπουν στο στόχαστρο. Γι' αυτό λοιπόν χρειαζόμαστε ένα μητρό με δημόσια πρόσβαση. Α, πότε το στόχος παρόλα αυτά θα πρέπει να είναι αυτό το οποίο τώρα ήταν ε, νόμιμο αλλά ανήθικο. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να τεθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στο παγκόσμιο επίπεδο προκειμένου να καταστούν παράνομε αυτές τι πρακτικές. Ευχαριστώ πολύ, λέει η πρόεδρο. Τώρα, από του συντηρητικού συνταρρυθμιστέ, ο κύριος Φωτίγκα έχει το λόγο. Η κυρία Φωτίγκα, συγγνώμη. Ευχαριστώ. Κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής, κυρίες και κύριοι, Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι όλες οι θετικές πρωτοβουλίες που περιγράφονται στο τελικό έγγραφο της διάσκεψης των G20. Στόχος είναι να φτάσουμε στην ανάπτυξη και τη δημιουργία ουσιαστικών θέσεων εργασίας. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Μας ενδιαφέρουν ε, τα προγράμματα υποδομών έτσι ώστε να προσαρμόσουμε τα τραπεζικά συστήματα και να προωθήσουμε τις ε, υποδομές, τις κομβικές υποδομές. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι και το θέμα της ασφάλειας που έχει και την οικονομική της διάσταση. Όταν εκλείπει δεν υπάρχει ανάπτυξη. Το θέμα αυτό όμως δεν αντικατοπτρίζεται στο έγγραφο των G20. Μετά από πρόσβαση των χωρών της Ευρώπης από όπου προέρχομαι εγώ στο ΝΑΤΟ, Είχαμε νέες άμεσες επενδύσεις στη χώρα μας, προωθήθηκε το πνεύμα του επιχειρήν, αλλά δυστυχώς υπήρξε μία μεγάλη απειλή στην περιοχή μας, η απειλή που προέρχεται από τις βαλκανικές χώρες. Και εσείς ως Κομισιόν και το Συμβούλιο δεν εκπροσωπήσατε, ε, παρά ένα, δεν εκπροσωπήσατε παρά ένα μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν μιλήσατε για αυτές τις απειλές κατά της περιοχής μας. γιατί φτάσαμε συμπεράσματα όπως τα ήθελε ο Βλαμιντίμιρ Πούτιν ε, εξ Φιλελευθέρων, ο κύριος ε, Τσίτς έχει το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Αυτό που μας ε, ενδιαφέρει είναι η ανεργία των νέων, κυρίως το 75, τα 75 εκατομμύρια είναι νέοι Παγκοσμίω στο Brisbane ε, προβήκαμε στην ανάλυση της κατάστασης που είναι σαφής. Ίσως ε, και τα στοιχεία υπερβαίνουν αυτά που χορηγήθηκαν. Έγινε λόγος για την ανάγκη να βρεθεί εργασία για τους νέους. Έγινε λόγος περισσότερες φορές ε, για το θέμα αυτό. και για την ισότητα δικαιωμάτων μεταξύ ανδρών και γυναικών. Οι γυναίκες θα πρέπει να έχουν ίσα δικαιώματα όσον αφορά την πρόσληψη και την απασχόληση. Σε παγκόσμιο επίθετο, επίπεδο θα πρέπει να υπάρχει ανάπτυξη για να βγούμε από την κρίση. Σήμερα αναμένουμε μαζική συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων για επενδύσεις σε μεγάλα προγράμματα και οι ΜΜΕ δημιουργούν ανάπτυξη. Θα πρέπει να μιλήσουμε και για τις κλιματικές αλλαγές και για την πράσινη οικονομία και για το πράσινο ταμείο, καθώς και την πράσινη βιομηχανία. Χρειάζονται εταιρικές ε, οικονομικές σχέσεις όπου να συνδράμουν και ο ιδιωτικός και ο, ειδικός, ο δημόσιος τομέας. διότι διακυβεύονται πολλά χρήματα και πολλές φορές δεν ε, φορολογούνται τα χρήματα εκεί όπου παράγονται. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Φερέιρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τα αποτελέσματα των G20 δείχνουν την εμβάθυνση μιας κρίσης. Δυστυχώς οι μεγάλες καπιταλιστικές δυνάμεις δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τους συστημικούς κινδύνους. Επειδή πρόκειται για συστημική κρίση, δεν θα βρεθεί λύση παρά μόνο αν ε, ξεφύγουμε από αυτό το άδικο σύστημα. Μέσα στα πλαίσια της στασιμότητας πολλών οικονομιών στην Ευρώπη υπάρχουν χιλιάδες μέτρα για την ε, ανάπτυξη της οικονομίας που δεν οδηγούν πουθενά. Θα πρέπει να εφαρμόσουμε την ε, συνταγή του Keynes έτσι ώστε να μην, δίνονται, να μην δίνεται δημόσιο χρήμα στις πολυεθνικές. Μιλάμε για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, αλλά δεν έγινε λόγος για τους φορολογικούς παραδείσους και για την απορρίθμιση του οικονομικού συστήματος καθώς και άλλες εγκληματικές δράσεις όπως το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος. Σας ευχαριστώ από την ομάδα του EFTD. Ο κύριος Μάχ για δύο λεπτά έχει το λόγο. Ο κύριος Φερέρα δεν τελείωσε αυτό που ανέφερε, αλλά θα συνεχίσω εγώ στο σημείο αυτό. Δεν σας φαίνεται υποκριτικό ότι λέμε ότι τα κέρδη θα πρέπει να φορολογούνται εκεί που πραγματοποιούνται και εκ παραλλήλου έχουμε τον κύριο Γιούνκερ υπεύθυνο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Πρωθυπουργό μιας χώρας η οποία ήταν και είναι φορολογικός παράδεισος προσφέροντας μεγάλες φορολογικές ελαφρύνσεις στη χώρα του. Μιλήσατε για το εμπόριο. Συμφωνώ ότι το ελεύθερο εμπόριο μπορεί να υποστηρίξει την ανάπτυξη, αλλά δεν σας φαίνεται υποκριτικό το γεγονός ότι διαπραγματευόμαστε μια εμπορική συμφωνία με τη ΣΥΠΑ που περιλαμβάνει μια ρήτρα διαιτησία. Και παράλληλα μιλάμε για την γέρεση της εταιρεία Google όταν μιλάμε για το TTIP, τη συμφωνία TTIP, νομίζω δεν θα είναι η πρώτη η περίπτωση διατησία όπου οι Ευρωπαίοι Φρολογούμενοι θα κληθούν να πληρώσουν τις ε, ΕΠΑ. Μιλήσατε για τις επενδύσεις και πόσο σημαντικό είναι. Σύμφωνο. Αλλά και πάλι η λύση που προσφέρεται είναι υποκριτική. Ο πρόεδρος Γιούνκερ έχει υποβάλει μία ιδέα την οποία σύμφωνα με την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πάρει 80 δισεκατομμύρια, θα προσθέσει 5 δισεκατομμύρια και η ΕΚΤ και αυτά θα βγουν με κάποιο θεματουργό τρόπο σε 325 δισεκατομμύρια. Δεν σας φαίνεται και αυτό υποκριτικό. Μιλάτε για ανάπτυξη, μιλάτε για θέσεις απασχόλησης, αλλά εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουμε ούτε ανάπτυξη ούτε θέσεις απασχόλησης τη συνθήκη της Λισαβόνας είχαμε, τη στρατηγική της Λισαβόνας είχαμε μέχρι το 2010 για να καταστούμε η πιο ανταγωνιστική οικονομία στον κόσμο, αλλά τελικά είμαστε μια οικονομία που δεν αναπτύσσεται καθόλου. Τουλάχιστον αυτό, αυτό παραταχθείτε στον εαυτό σας. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Ο κύριος Μπέι για ένα λεπτό παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, πέρα από το μηντιακό θέαμα, δεν Υπήρχαν και πολλά να περιμένει κανείς από αυτή τη νέα έκδοση του G20, εκτός από την επιβεβαίωση του προσανατολισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία υποδουλώνεται όλο και περισσότερο στην ιδεολογία της παγκοσμιοποίησης και στα συμφέροντα των ΗΠΑ. Ενώ ορισμένοι συνεχίζουν να εμένουν στο όνειρο μιας παγκόσμιας κυβέρνησης υπό αμερικανικό προτεκτοράτο, όλοι, όπως και η Ρωσία, η οποία δεν είναι καθόλου απομονωμένη όπως νομίζετε, ετοιμάζουν αυτόν τον ε, κόσμο με διαφορετικούς πόλους όπου υποτίθεται οι πατριώτες όλων των χωρών ε, αυτό επιθυμούν. Εκτός από τις αντιρωσικές κορώνες του Αυστραλού Πρωθυπουργού είχαμε και την συλλογική ιστερία της, Ευρω... ιστερία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλό το Κοινοβούλιο να εμπνευστεί από τη μεταναστευτική πολιτική της Αυστραλίας η οποία είναι σαφέστατη. Ε, η επιχείρηση του Σεπτεμβρίου του 2013 κυρίαρχα σύνορα ουσιαστικά κατάφερε να αποτρέψει ε, τους υποψήφιους μετανάστες να, από το να έρθουν στην Αυστραλία και στέρεψε το δίκτυο των διακινητών. Μπορούμε και εμείς να κάνουμε το ίδιο έτσι ώστε να μην βρίσκουν το θάνατο όσοι θέλουν να πλησιάσουν δυστυχώς τα σύνορά μας. Μπορούμε να έχουμε λοιπόν αποτελεσματική μεταναστευτική πολιτική. Κυρία Σπυράκη, για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η δέσμευση των G20 να εργαστούν για τόνωση της ανάπτυξης και της οικονομικής ανθεκτικότητας είναι πλέον άκρος επίκαιρη και είναι επίκαιρη όχι γιατί μόνο η ανάπτυξη παγκοσμίω αλλά και στην ευρώπη είναι πολύ ασθενή, ασθενέστερη πάντω από την αναμενόμενη αλλά και γιατί λίγες ώρες πριν ο πρόεδρος Γιούγκερ παρουσίασε εδώ το επενδυτικό σχέδιο των 315 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ευρώπη. είναι ένα σχέδιο φιλόδοξο που αν πετύχει έχει τη δυνατότητα να πετύχει το στόχο να δημιουργήσει δηλαδή περισσότερες από ένα εκατομμύριο νέες θέσεις εργασίας την επόμενη τριετία χωρίς ωστόσο να επιβαρύνει την ευρώπη με χρέος. είναι ένα σχέδιο βεβαίως το οποίο θα πρέπει να μας διευκρινιστεί λεπτομερώς και οι λεπτομέρειες έχουν σημασία καμιά φορά ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. πρέπει δηλαδή να μας πούνε από την ευρωπαϊκή επιτροπή πώς προκύπτουν τα 315 δισεκατομμύρια ευρώ, καθώς ο πολλαπλασιαστής είναι άκρος φιλόδοξος, φτάνει το 15 μέσω της μόχλευσης των κεφαλαίων. Ένα ακόμη σημαντικότερο ερώτημα είναι τι θα γίνει με τις χώρες που βρίσκονται σε κρίση. Ο πρόεδρος Γιούγκερ σήμερα είπε ότι οι χώρες που βρίσκονται σε κρίση έχουν προτεραιότητα. Η πρώτη χώρα που υπέστη πολύ μεγάλες επιπτώσεις από την κρίση είναι η Ελλάδα ποια θα είναι η διαδικασία ώστε οι χώρες αυτές να προηγηθούν στα προγράμματα που θα προέρχονται από το νέο ταμείο. αυτό που πρέπει να γίνει ωστόσο είναι να κρατήσουμε την πρωτοβουλία της επιτροπής γιατί είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία και έρχεται να απαντήσει αμέσως στη δέσμευση των g. 20 και επίσης πρέπει να μας δοθούν αμέσως διευκρινήσεις για το πώς θα κινηθούν από την επιτροπή και από την ευρωπαϊκή τράπεζα επενδύσεων σε σχέση με τα νέα καινοτόμα πλέον χρηματοδοτικά εργαλεία. Τι θα είναι αυτά. Είναι πολύ σημαντικό μέρος του νέου επενδυτικού σχεδίου και πρέπει να ξέρουμε. Να ξέρουμε όχι γιατί βλέπουμε αρνητικά την πρωτοβουλία της Επιτροπής. Να ξέρουμε για να οθήσουμε προς την κατεύθυνση του να υπάρχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη. Να περιοριστεί το ρίσκο. Είναι προφανές ότι το νέο σχέδιο έχει έναν πολύ βασικό, πολύ, πολύ φιλόδοξο αλλά και πολύ σπουδαίο στόχο. Να αλλάξει την εικόνα της Ευρώπης δεν έχουμε χρόνο στην ευρώπη αυτό αποτυπώθηκε στη διακήρυξη των g 20 δεν έχουμε χρόνο πολύ περισσότερο στις χώρες που υπέστησαν τις επιπτώσεις της κρίσης. σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Μιλάμε για ένα πολύ σημαντικό θέμα, αλλά θα ήθελα να τηρήσετε το χρόνο ομιλία σας, γιατί θα πρέπει να σεβαστούμε τους επόμενους ομιλητές. Ο κύριος Γκουτιέρες Φρέτ. Είναι ε, γεγονός ότι δεν είμαι υπέρμαχος των G20. Μετά από την πτώση των ε, Lehman Brothers, στην ουσία δεν γίνεται τίποτα. Δεν υπάρχει καλύτερη ρύθμιση των οικονομικών αγορών αλλά κύριε Επίτροπε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μίλησε για τον δίκτυο ανάπτυξη που είναι κοντά στο μηδέν. Ε, δίκτυ ανεργίας πολύ υψηλό κίνδυνο αποπληθωρισμού και μεγαλύτερη ευαλωτότητα των αγορών. Όλοι ζητούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αλλάξουμε. Μας ζητούν να κάνουμε περισσότερα πράγματα και πιο σημαντικά για να προωθήσουμε την ανάπτυξη. Πρόκειται για κοινή λογική. Αλλά εμεί ε, προβάλλουμε μία Ευρώπη διχασμένη. Υπάρχουν εκείνοι που παρετούνται και εκείνοι που προβάλλουν κίνητρα. Η νομισματική πολιτική, όσο διευρυμένη και να είναι, δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Χρειαζόμαστε περισσότερα κίνητρα δεν πρέπει να δεχτούμε την οικονομική λιτότητα όπως τη ζητάει η Γερμανία. Οι ε, μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να είναι σωστές, να ε, οδηγήσουν σε μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη. Χρειαζόμαστε περισσότερα ε, έσοδα να αποφύγουμε την φοροαποφυγή και την φοροδιαφυγή. Και τέλος χρειαζόμαστε οπωσδήποτε αλληλεγγύη για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κοινωνία που έχει παρετηθεί ακριβώς επειδή δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Ο κύριος Σίλικ, για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πρώτα, κύριε Επιτροπέ. Η σύνοδος του G20 ανέφερε και πάλι την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Δεν υπάρχει, μάλλον είναι Προκαλεί έκπληξη το γεγονός αυτό. Γιατί η Ευρώπη ξέρει ότι δεν θα υπάρξει ανάπτυξη γιατί αυξάνει τους φόρους, δημιουργεί όλο και πιο δύσκολο επιχειρηματικό κλίμα, θέτει μη ρεαλιστικούς στόχους και μετά όλοι ευνηδιάζονται από το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις φεύγουν από την Ευρώπη και δεν υπάρχει ανάπτυξη. Πιο πολλές δημόσιες δαπάνες χρειάζονται, λέτε πιο πολλά χρέη. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματικά θέλει να επιλύσει το πρόβλημα της οικονομικής ανάπτυξης και πραγματικά θέλει να μειώσει την ανεργία, θα πρέπει να αφήσει τις χώρες που δεν μπορούν να διαχειριστούν τα χρήματά τους να πτωχεύσουν, να σταματήσει να ρυθμίζει, να σταματήσει το μη ρεαλιστικό αυτό κλίμα και να βελτιώσει το περιβάλλον για τις επιχειρήσεις συστηματικά. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Επόμενος ο μελητής, ο κύριος Μαζουρι... Μαζουρώνης. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Συνάδελφοι, μπορούμε να χαρούμε διότι οι ηγέτες των μεγάλων δυνάμεων συναντήθηκαν στη σύνοδο του g 20 στο Πέιν και συζήτησαν για τα προβλήματα που ταλανίζουν το πλανήτη μας και χαίρομαι που συζήτησαν για την κλιματική αλλαγή, για την αηφόρο ανάπτυξη μεταξύ άλλων. Οφείλω να πω ότι οι ηγέτες ε, του κόσμου ένωσαν τις δυνάμεις τους έναντι της ρωσικής απειλής. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν παρέστη στη σύνοδο του G20, αλλά τα περισσότερα μέλη ξεκάθαρα του είπαν ποια είναι η γνώμη τους για την κρίση και την κατάσταση στην Ουκρανία. Και χαίρομαι ιδιαίτερος διότι θα οφείλει να το λάβει αυτό υπόψη του, ε, προσπαθώντας να βρούμε μια ειρηνική λύση. Πρέπει να δούμε και τι γίνεται στα ρωσο-λιθουανικά σύνορα. Θα πρέπει η Ρωσία να συνέλθει και να κάνει πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά που πρέπει. Ευχαριστώ, κύριος Βιλίνσκι, για 1,5 λεπτό. Σας ευχαριστώ πολύ κυρίες και κύριοι. Να φανταστούμε ότι η κοινότητα των 20 πιο πλούσιων χωρών είναι μια πολύ σημαντική παρτίδα του κόσμου. Δύο τρίτα του εμπορίου αντιπροσωπούν και σε ό,τι αφορά το ΑΕΠ και όταν ε, συνέρχεται λοιπόν μια τόσο σημαντική και δυνατή ομάδα περιμένω και σημαντικές λύσεις και δεν περιμένω λοιπόν ε, τον κύριο Γιούγκερ να μας ε, κάνει παρεδόση. Περιμένουμε νέα χρήματα. Από την κρίση του 2008 θα πρέπει να γίνει, ε, μετά την κρίση του 2008 θα πρέπει να γίνει διαχωρισμός των τραπεζών και των επενδύσεων για να μην παίζουν καζίνο χρηματοδοτικό, αλλά να έχουν υποχρεώσεις σε ό,τι αφορά τις επενδυτικές τράπεζες για να υπάρξει διάκριση προκειμένου να υπάρχει σταθερότητα στα οικονομικά και κατά δεύτερον σε ό,τι αφορά τις συναλλαγές εκτός χρηματοστηρίου να ρυθμιστούν σε ό,τι αφορά τα over-the-counters. Δύο τρίτα όλων των ε, διευθυντών αφήνουν τις τράπεζες ελεύθερες και όλο πιο μεγάλες είναι οι δομές που δεν ελέγχονται, που δεν ρυθμίζονται και ήταν μεγάλο το κενό μεταξύ των G7 και των BRIC από την άλλη. Αυτό το κενό, αυτό το χάσμα όλο και διωγγώνεται, όλο και οξύνεται. Δεν χρειάζεται λοιπόν αυτό, χρειαζόμαστε να εξυπηρετούν αυτές οι μεγάλες δυνάμεις το συμφέρον των άνθρωπων και να μην αφήνουμε έτσι τις ε, χρηματοοικονομικές αγοράς πλέον. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπάλλας, 1,5 λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, η ΕΚΤ, ο, ο ΣΑ, το και τώρα η G20 λένε ότι όλες οι προϋποθέσεις που είχαμε ε, στον οικονομικό τομέα ήταν νεοφιλελεύθερης η ε, φύση και δεν λειτουργούν πλέον. Σήμερα θα πρέπει να αυξήσουμε τη ζήτηση σε διεθνές επίπεδο για τα αγαθά και τις υπηρεσίες. Και γι' αυτό γνωρίζουμε ότι το θέμα της φοροδιαφυγής και της φορολογικής απάτης πρέπει να αντιμετωπιστούν. Ξέρουμε το, ότι το θέμα της οικολογικής ε, αντιμετώπισης είναι κάτι το σωστό. Ο Συνάδος το τόνισε αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να λάβουν υπόψη αυτά, αυτό ακριβώς σαν πρόκριμα, να αντιμετωπίσουμε τη φόρο διαφυγή και να πάμε πολύ πιο μακριά ως προς το σχέδιο επενδύσεων, σήμερα το πρωί αναφέρθηκε το πρώτο βήμα να γίνει στοχοθέτηση των επενδύσεων έτσι ώστε να υπάρξει αυτή η, αυτός ο οικολογικός ε, μετασχηματισμός και να είμαστε πρωτοπόροι. Θα πρέπει να αλλάξει η οικονομική μας πολιτική, ακόμα και οι G20 το λένε. Είναι καιρός να ακολουθήσουμε αυτή την οδό. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Μποστινάρου για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε, η ομάδα των σοσιαλιστών και δημοκρατών γνωρίζουν τα μικρά αυτά βήματα που έγιναν από τους G20 έτσι ώστε να αυξηθεί το ΑΕΠ κατά 2% τουλάχιστον. Όμως ε, Εάν άλλα κράτη καταφέρουν να αντιμετωπίσουν την ε, κρίση ενώ η Ευρώπη όχι, ε, δεν σημαίνει ότι οι άλλοι είχαν την καλύτερη συνταγή. Θα πρέπει να αναπτύξουμε τις επενδύσεις και τις ε, θέσεις εργασίας όπως αναφέρθηκε σήμερα στο Κοινοβούλιο. Επίσης θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την φοροδιαφυγή την διασυνοριακή με ανταλλαγή πληροφοριών. Τα κέρδη θα πρέπει να φορολογούνται εκεί που παράγονται. Ας το αναγνωρίσουμε αυτό. Αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα. Γιατί γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν φτάνουμε στο έπτον είπα έγινε λόγος για τις κλιματικές αλλαγές. Εμείς όμως οι Ευρωπαίοι δεν δέχτηκαμε το μεγάλο deal που έγινε μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ. Δεν έγινε λόγος για το έμπολα. Δεν το αναγνωρίζει το G20. Τα κράτη δεν κατάφεραν να προβλέψουν την κρίση ή να την θεραπεύσουν. Δεν θα πρέπει να μεγεθυνθεί και να φτάσει σε ένα δυσβάστακτο οικονομικό και κοινωνικό κόστος. Αυτός είναι και ο ρόλος, ο ηγετικός ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα πρέπει να εισακουστεί. Ευχαριστούμε ο κύριος ε, David Μάρτιν για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρε, τέσσερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μέλη και του G20 και δυστυχώς για όλους εμάς η ανάπτυξή μας έχει φτάσει σε τέλμα σε σχέση με τις υπόλοιπες 16 χώρες του G20, όπου, των οποίων η ανάπτυξη πραγματικά ανθεί. Καλωσορίζω τα επενδυτικά σχέδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το εναρκτήριο επιτέλους λάκτισμα στην ευρωπαϊκή οικονομία. Ωστόσο, δεν μπορούμε να έχουμε ε, αηφόρο οικονομική ανάκαμψη μέσω δανείων μόνον. Θα πρέπει να μπορέσουμε να έχουμε ανάπτυξη και να μπορέσουμε να έχουμε βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, να έχουμε σαφή ατζέντα. Είμαστε η μεγαλύτερη αγορά στον κόσμο. Δεν έχουμε συνειδητοποιήσει το δυναμικό μας. Το G20 επιβεβαίωσε ότι θέλει να μεταρρυθμίσει το πολυμερές ε, σύστημα εμπορίας και εγώ χαίρομαι γι' αυτό και χαίρομαι διότι ε, θα δοθεί συνέχεια σε όλα αυτά τα πράγματα. Όμως ε, ε, δυστυχώς οι πολυμερείς ε, συμφωνίες δεν θα φανούν άμεσα στον ορίζοντα. Θα πρέπει να προχωρήσουμε και τις διμερείς συμφωνίες. Π.χ. αυτή με την Σιγκαπούρη να κυρωθεί. Ε, θα πρέπει να πετύχουμε στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία. Να έχουμε σωστή και καλή επενδυτική συμφωνία με την Κίνα. Όχι με οποιοδήποτε τίμημα, αλλά με ένα επαρκές και ικανοποιητικό τίμημα βάσει αυτών που συμφωνήθηκαν στο G20 και θα πρέπει οι συμφωνίες αυτές να τονίζουν τη δίκαιη ανάπτυξη, την αηφόρα ανάπτυξη, τις δίκαιες συνθήκες εργασίας, τη φορολογική διαφάνεια και τη ε, σωστή κανονιστική πλαισίωση. Εάν τα πετύχουμε αυτά στις διμερείς μα συμφωνίες, θα συμβάλλουμε στους στόχους του G20 και θα καταφέρουμε να επεκτείνουμε την ευρωπαϊκή οικονομία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κι εγώ. Επόμενος ομιλητής, κύριος Ντάντι. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε συνάδελφοι. Η διάσκεψη κορυφής του Brisbane προσπάθησε να δώσει μία απάντηση στην οικονομική κρίση που ζούμε. Η ανάπτυξη γενικότερα δεν αποτελεί μέλημα μίας χώρας, αλλά της παγκόσμιας κακέρας. Ο κύριος Γιούνκερ μας παρουσίασε ένα επενδυτικό σχέδιο που έχει τα όρια του βεβαίως, αλλά αποτελεί ε, μία κρίσιμη καμπή, διότι εγκαταλείπουμε το παλιό μονοπάτι της ε, λιτότητας. Θα πρέπει να κρατήσει επιθετική στάση η Ευρώπη ανά τον κόσμο και να είναι πρωταγωνιστής στις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις θα πρέπει να μετασχηματίσουμε αυτή την γυραλέα Ευρώπη και την κουρασμένη Ευρώπη σε ένα πρωταγωνιστή, όπως είπε χτες το σώμα αυτό ο Πάπας. Γιατί αυτό αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία για τις μελλοντικές γενναίες. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα μπαίνουμε στην διαδικασία Catch the Eye. Ο κύριος ε, Νίκολα Καπούτα έχει το λόγο πρώτος. Στη διάσκεψη του Brisbane μιλήσαμε για το ΑΕΠ, για τις νομισματικές αρχές, για το οικονομικό σύστημα, για τις διαρθρωτικές ε, μεταρρυθμίσεις. Όμως το τελικό ανακοινωθέν δεν αναφέρεται στους παραγωγικούς τομείς που ορίζουν την οικονομία Μιλώ για τις ΜΜΕ που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της Ευρώπης και κάθε μέρα προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την οικονομική συγκυρία, τη χειρότερη που ε, ζούμε μετά τον πόλεμο. Οι G20 θα έπρεπε να είχαν προβάλει προτάσεις και στο θέμα των φορολογικών παραδείσων. Ως προς το πρόγραμμα κατά της ε, διαφθοράς, θα δώσει καλύτερη διαφάνεια και στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα για να βελτιώσουμε και τις κλιματικές συνθήκες και να αντιμετωπίσουμε και την ανεργία των νέων που έχει φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Άτρετς. Thank you. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο κύριος Γκόζη είπε ότι τα αποτελέσματα του G20 ήταν ε, ε, θετικά σε ό,τι αφορά την αντίληψή του στην οικονομία. Αν αυτό αποτυπώνει αυτά που είπε ο κύριος Γιούγκερ σήμερα το πρωί σε ό,τι αφορά αυτό το τεράστιο ποσό ε, ευρωπαϊκής χρηματοδότησης το οποίο θα σπαταλήσει πάνω σε μια οικονομία η οποία ήδη έχει χρεωθεί 90% του ΑΕΠ της και το 50% του ΑΕΠ της θα διατηθεί μόνο κακοδιαχείριση και απελπισία θα προκαλέσει αυτό το πρόγραμμα και πραγματικά αν αυτό αποτελεί το σκοπό μας να μας βοηθήσει ο Θεός. Σας ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Και τώρα να δώσω το λόγο στον Επιτροπό για να απαντήσει στα θέματα τα οποία ετέθησαν. Ο κ. Δομπρόφσκης. Ε, Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη συζήτηση, για τα σχόλιά σας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει όλες σας τις παρατηρήσεις και θα τις αξιοποιήσει καταλήλως, καθώς και τις συστάσεις σας καθώς ξεκινάει η ε, τουρκική προεδρία του G20 στη συνέχεια αυτής της χρονιάς και της επόμενες. Είμαι βεπισμένος ότι το G20 είναι ένας θεσμός ο οποίος θα παραμείνει, διότι είναι ένα φόρουμ όπου συναντιόνται οι ανεπτυγμένες και οι αναδυόμενες χώρες και μπορεί πραγματικά να οδηγήσει τις οικονομίες σε οδούς πιο ασφαλείς έξω από την κρίση. γνωρίζουμε και από δική μας εμπειρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι ο δρόμος είναι δύσκολος, ότι θα πρέπει να σημειωθεί πρόοδος σε παγκόσμιο επίπεδο έτσι ώστε να έχουμε ε, σημαντική βελτίωση στις ε, κατατόπου ε, περιφέρειες ανά τον κόσμο. Πολλά ήταν τα παραδοτέα στο G20 με το ανακοινωθέν πιστεύουμε πραγματικά ότι θα ενισχυθεί η ανάκαμψη της οικονομίας στην Ευρώπη. Ο πολλοί ομιλητές αναφέρθηκαν στην ασφάλεια σε σχέση με την κατάσταση στην Ουκρανία. Παρόλο που επισήμως αυτό δεν αποτέλεσε μέρος της ημερήσιας διάταξης του G20, συζητήθηκε εκτεταμένα στο περιθώριο της συνόδου του G20 και άλλωστε ο πρόεδρος Γιούνκερ είχε μια σοβαρή ε, συζήτηση για το θέμα αυτό με τον πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, τον κύριο Βλαντιμίρ Πούτιν, ως προς το G20. Το 2015 θα πρέπει να είναι το έτος όπου θα εφαρμοστεί και θα ολοκληρωθεί η ημερήσια διάταξη, η εφαρμογή όλων αυτών για τον οποίο, τα οποία συζητιόνται. Μιλούμε για την ανάπτυξη και την ανάκαμψη των οικονομιών και αυτό θα είναι μέρος της ημερήσιας διάταξης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον Επίτροπο κ. Ντομπρόφσκιφς. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Γκόζη ε, που εκπροσωπεί το Συμβούλιο. Παρακαλώ. Θα ήθελα να αναφερθώ στην ανάγκη αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής. Θα πρέπει να γίνει και σε επίπεδο G20, αλλά και με βάση τη νέα μας νομοθεσία να καταπολεμήσουμε τους φορολογικούς ε, παραδείσους σε παγκόσμιο επίπεδο και να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ακριβώς ε, προβάλλουμε σαν έργο κατά τη διάρκεια της προεδρίας μας επίσης ε, θα πρέπει να συμφωνήσουμε ως προσυνεργασία συνεργασία μεταξύ δημόσιων διοικήσεων. Ο συνάδελφος Μαρτίν μίλησε για την ανάγκη προώθησης της εμπορικής ατζέντα σε πολυετές επίπεδο και στους G20 τα κράτη θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να φτάσουμε στη συμφωνία ως προς το TTIP. έγιναν σοβαρά βήματα φτάνοντας στο στόχο της ε, εμπορικής συμφωνίας ε, μέσω ΓΚΑΤ, μέσω Σιγκαπούρης και Ιαπωνίας, όπως υπενθύμησε ο συνάδελφος ε, Σάιμον. Σεφκοβιτς αναφέρθηκε στα αριθμητικά στοιχεία που υπενθυμίσαμε, γιατί αυτό είναι το σημείο αναφοράς από το οποίο απορρέει οποιαδήποτε οικονομική και κοινωνική πρόταση. 200 εκατομμύρια άνεργοι σε παγκόσμιο επίπεδο χρειάζονται απαντήσεις για να συμμετέχουν οι πάντες στην αγορά εργασίας. Αυτό το θίξαμε και σε επίπεδο G20, προώθηση του επιχειρήν. Να βοηθήσουμε εκείνους που είναι πιο ευάλωτοι, που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες. Αυτό θα πρέπει να μας αποσχολήσει ιδιαίτερα. Επίσης θα πρέπει να προωθήσουμε τις ε, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας Τέλος, ε, η Μπάλας Ντάντε Γκουτιέρες Πριέτο μίλησαν για την ανάγκη την οποία συμμεριζόμαστε μία αλλαγή της παγκόσμιας οικονομικής πολιτικής και στους G20. Λάβαμε πολλά μηνύματα ως Ευρωπαϊκή Ένωση για να αλλάξουμε την ταχύτητά μας. Κάτε μας, αυτό αποτελεί ένα βασικό μήνυμα. Βεβαίως χρειάζονται νέα οικονομικά κίνητρα να εκμεταλλευτούμε κάθε ευελιξία στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και στην στρατηγική ατζέντα μας. Αυτό είναι το σημείο εκκίνησης, το οποίο βρήκαμε και στο πρόγραμμα Juncker και τα λόγια του μαζί με τον Αντιπρόεδρο Κατάινεν που μίλησαν για την εθνική συνεισφορά η οποία θα είναι ουδέτερη σε σχέση με το ε, σχέδιο σταθερότητας και ανάπτυξης. Βεβαίως, οι δημόσιες δαπάνες που θα γίνουν υπέρ των επενδύσεων ε, δεν θα πρέπει να θεωρηθούν τρέχουσες δαπάνες. Είδαμε τη σωστή εφαρμογή αυτού του πλαισίου με βάση το σχέδιο Juncker και πιστεύουμε ότι εάν εφαρμοστούν αυτοί οι κανόνες θα επεκταθούν και σε άλλα επενδυτικά μέσα που έχουμε μέσω των περιφερειακών συγχρηματοδοτήσεων και της πολιτικής συνοχής για τους αναπτυξιακούς στόχους που θα πρέπει να θεωρηθούν ουδέτερη δύναμη του Συμφώνου Σταθερότητας. Μιλήσατε για την αλληλεγγύη. Χρειάζεται μεγάλη αλληλεγγύη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφέρθηκε, αναφέρεται σε 21 άρθρα των συνθήκων. Είδαμε ότι είμαστε πεπισμένοι για την χρήση της αλληλεγγύης σε διάφορους ε, τομείς Ελπίζουμε αυτή να είναι μία δέσμευση που θα υλοποιήσουν τα τρία θεσμικά όργανα στη Νέα Θητεία. Ο, ο κύριος Έθερης μίλησε για την επίκληση στο Θεό. Βεβαίως μπορούμε να επικαλεστούμε το Θεό, τον οποίο επικαλέστηκε χτες και ο Πάπας και ίσως μας εμπνέει, αλλά δεν νομίζω ότι έτσι θα ανταποκριθούμε στην ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας που απαιτούν οι πολίτες μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ λεπτομερή αυτή απάντηση από πλευρά της Προεδρίας για τα σχόλια που έγιναν κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Και τώρα λοιπόν ολοκληρώθηκε η συζήτηση αυτή και θα περάσουμε κατευθείαν στο επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη που είναι η δήλωση της Επιτροπής ότι αφορά την ενιαία ψηφιακή αγορά. Τρεις, ε, τρία σχέδια ψηφίσματος είχαμε από το ΕΛΚ και τους Σοσιαλδημοκράτες